τελευταίο σημείο η Βόρεια Κορέα. Ξεκινώ με τους εισηγητές παραβιάζεται εντελώς τους κανόνες από τους 751 έχουμε καμιά 45 βουλευτές. Για διαφωτίστε σας παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς που μπαίνουμε στον κόπο να παραμείνουμε εδώ. Γιατί δεν μας δίνετε το λόγο στο πλαίσιο της αντικασίας τιάει; Και αν αποφασίσετε, και δεν ποτέ να μην μας δώσετε τελικά το λόγο. Από απλή ε, συναδελφικότητα. Δεν θα έπρεπε να μας πείτε γιατί, με τι, πού βασίζεστε και δεν μας δείτε το λόγο. Απάντηση. Ακούστε. Νομίζω ότι είμαι ο πρόεδρος που κάνει περισσότερες προσπάθειες από τους υπολείπους ίσως προέδρους για να δίνω το λόγο σε όλους. Έχετε πάρει το λόγο πολλές φορές σήμερα, δεν σας είδα, σας το συγγνώμη τη συγκεκριμένη φορά. Βέβαια, αυτό δεν έχει να κάνει τη δική μου προσωπική ε, βούληση και ποτέ νομίζω δεν ε, ε, υποστήκατε άδικη μεταχείριση από εμένα. Ο κύριος Σκλέτσκ. Έχει το λόγο για δύο λεπτά. Господин gospodine Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Μπορείτε παρακαλώ να με προσέξετε. Κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι εδώ ο κύριος Σκρέλτς. Okay, thank you. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σημαντική η πληροφορία αυτή. Αφού δεν είναι εδώ λοιπόν, θα δώσω τώρα στην κυρία Ντινόλφη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ζητώ συγγνώμη εκ μερού του εισηγητή συντάκτη που δεν μπορεί να είναι εδώ. Μόνο και μόνο πυρηνικά η λέξη αυτή με κάνει να ρηθιώ. Δεν μπορούμε να μιλάμε για την περίπτωση των πυρηνικών ε, χωρίς να μην βλέπουμε πόσο αμφιλεγόμενο είναι το θέμα. Πρέπει και εμείς στην Ευρώπη να διαλύσουμε την πυρηνική μας διοργάνωση και να πάρουμε τις σχέσεις με χώρες που προκαλούν. Είναι καλό παράδειγμα εδώ πως ε, η Βόρεια Κορέα για το πώς μπορούμε να είμαστε δίκαιοι. Η πρόσφατη είδηση ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε αποφάσισαν να ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού του πυρηνικού του εξοπλισμού και το πρόγραμμα αυτό θα ε, περιλαμβάνει και την Ιταλία με 70 ατομικές βόμβες που θα ε, που είναι βόμβες νέα γενιάς και οι οποίες καταστρέφουν και το υπέδαφος, πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο να έχουμε το δικαίωμα να δακτυλοδεικτούμε το καθεστώς της Βόρειας Κορέας και να σκεφτούμε ότι η οποιαδήποτε αντιπαράθεση μεταξύ κρατών μελών ή με τρίτες χώρες θα έπρεπε να ξεκινάει από τις ΗΠΑ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντέβα. μισή λεπτό. Πρόεδρε, Μιλώ ως πρόεδρος αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Κορεατική Χερσόνησο. Και είναι πολύ δύσκολο να σηκώνομαι σήμερα το απόγευμα και να μιλώ για όσα γίνονται στην Βόρεια Κορέα. Είναι πολύ κρίμα όταν ακούμε ότι έγινε μια πυρηνική δοκιμία από το Βόρειο Κορεϊκό καθεστώ. Το Ευρωκοινοβούλιο και την προσωπία μου είχαν εργαστεί σκληρά, ε, ε, ε εξαιρετικά σκληρά τα τελευταία χρόνια, για να ε, συσφιχθούν οι σχέσει Βορρά και Νότου στην Κορεατική Χεξόνησο. Προσκληθήκαμε μάλιστα και από τι δύο πλευρέ ώστε να συντάξουμε μια συνθήκη ειρήνευση που αυτή τη στιγμή ε, δεν θα μπορούσε να επίσταται με την έλλειψη σχέσεων ε, μεταξύ Βορρά και Νότου. Ο διαχωρισμός ε, είναι ένας διαχωρισμός που έχει ξεκινήσει από δεκαετίες. Θα μπορούσε να υπάρξει μια εκεχηρία όπως έχει συμφωνηθεί, αλλά αυτό δεν είναι συνθήκη ειρήνευσης. Θα έπρεπε λοιπόν με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Κίνας, ε, της Ρωσίας και όλων των ενδιαφερομένων εταίρων να καταλήξουμε σε ένα θετικότερο αποτέλεσμα. Θέλουμε οι σχέσεις μας και ο διάλογος να διατηρηθεί με την ε, Βόρεια Κορέα, ακόμη και αν παίζουν ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι. Ε, δεν έχει κανένα νόημα έτσι κι αλλιώς, εάν το δει κανεί ούτε για τους ίδιους, ούτε για την διεθνή ειρήνη. Δεν μπορούν να δημιουργήσουν οικονομικές δομές ε, κατασκευάζοντας πυρηνικά. Ε, όταν ε, οι πολίτες τους πεινάνε και η οικονομία τους ε, φθήνει. Θα πρέπει λοιπόν να αφήσουμε τις πόρτες μας ανοιχτές και εγώ από πλευράς μου αυτό σκοπεύω να κάνω. Mr. Δέχεστε γαλάζια κάρτα, παρακαλώ, την Γκραπίνη. Κύριε Ντέβα, βεβαίως. Παρακαλώ, κυρία Γκραπίνη, το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντέμβο, γνωρίζετε και, ε, ε, ήσασταν και εσείς μαζί στο ΡΙΑΝΤ ότι πρέπει ε, να βοηθήσουμε και εμείς για τη συμφιλίωση των δύο χωρών της Κορετικής κερσονήσου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως μπορεί να επηρεάσει αυτή τη διαδικασία. Γιατί ο Υπουργό Συμφιλίωση ε, τη Νότια Κορέα δεν μου φάνηκε να έχει ένα πολύ ε, συνοκτικό πρόγραμμα. Κύριε Γκραπίνη, είναι η απάντηση. Πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σα και αν δείτε όλου του συνομιλητέ μα σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Εμεί είμαστε οι μόνοι, μιλάω για την Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν έχει κάποια συγκεκριμένη, κάποιους συγκεκριμένους στόχους. Εμείς θέλουμε συμφιλίωση, θέλουμε ειρήνη, τελεία και παύλα. Και θέλουμε αυτό να το καταλάβουν οι Κινέζοι, οι Άπωνες, οι Βορειοκορεάτες, οι Νοτιοκορεάτες, οι ΙΠΑ. Και μόνο έτσι θα πετύχουμε πρόοδο, αν το κατανοήσουν όλοι οι υπόλοιποι. Άρα εμείς έχουμε μια μοναδική θέση και ένα μοναδικό ρόλο να διαδραματίσουμε. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Πρέντα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση για τη Βόρεια Κορέα είναι πολύ σημαντική για πολλούς και διαφόρους λόγους. Πρώτον, εντάσσεται στο κίνημα ε, καταγγελίας των πυρηνικών δοκιμών ε, της ε, Βόρειας Κορέας για τι οποίε περηφανεύεται ενώ κατά φορά παραβιάζει όλους τους κανόνες και αποσταθεροποιεί τη Χερσόνησο. Πρώτος λόγος αυτός. Δεύτερος, ένας Κορεάτης ήταν Υποψήφιο για το βραβείο Ζαχάρο φέτο, σε δεσμότατος Γιούν. Επίσημω όμως, επειδή δεν υπήρξε αρκετή υποστήριξη, δεν ήταν σε του επίσημου ε, υποψηφίου. Αλλά θα ήταν πολύ σημαντικό αν είχε γίνει αυτό. Γιατί το βραβείο Ζαχάροφ ε, έχει εγνωσμένη αξία και προβολή. Θα μπορούσε λοιπόν να βοηθήσει να βελτιωθούν ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, να υπάρξει μεγαλύτερη δεσμεύση. Γι' αυτό και δράτω με τι ευκαιρίε για να καλέσω όσου συναδέλφου θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν την Βόρεια Κορέα να υποστηρίξουν ε, για φέτο αυτή την υποψηφιότητα, γιατί κανένα Βορειοκορεάτη ούτε καν επίσημα δεν είχε οριστεί ω υποψήφιο για το βραβείο Ζαχάροφ. Ε, παρόλα αυτά πρόκειται για μια πολιταρχική χώρα. Και έχουμε δώσει σε άλλε σημαντικέ προσωπικότητε που ανήκουν σε απολυταρχικές χώρες, το βραβείο Ζαχάροφ. Ας κάνουμε αυτή την προσπάθεια φέτος λοιπόν. Να πω τώρα για τη Βόρεια Κορέα ότι η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει προτεραιότητα για την εξωτερική πολιτική και με αυτήν την έννοια στο ψήφισμά μας ε, καλούμε την κυρία Μαγκερίνη να παρακολουθεί την κατάσταση σε αυτή τη χώρα, εκ του σύνεγγης μάλιστα και να ε, ασκεί σταθερή πίεση. Θα ήθελα να ξαναμπεί ε, η Βόρεια Κορέα ε, στα θεματολόγια των ψήφισμάτων μας. Διότι είμαι αισιόδοξο. Πιστεύω ότι έχει δυνατότητα να αλλάξει χώρα και αξίζει ο ίδιος ο λαός της χώρας. Εμείς να είμαστε ε, προσιλωμένοι γιατί το καθεστώς δεν πρόκειται από μόνο του να πάρει κάποια πρωτοβουλία. διεθνής κοινότητα μόνο μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό το παράθυρο ευκαιρίας. Ευχαριστώ τώρα λόγο. Οι πυρηνικές δοκιμές που έκανε η Βόρεια Κορέα ήδη από τον Ιανουάριο καταδικάστηκαν από το, από το Συμβούλιο Ασφαλείας και εμείς καταδικάζουμε την άμεση απειλή κατά της ασφάλειας και της ειρήνης. Περαιτέρω <clears throat> προκλήσεις θα πρέπει να αποφευθούν με κάθε τρόπο με το να σταματήσει η Κορέα το πυρηνικό της πρόγραμμα και το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων. Θα πρέπει να βρεθεί μία λύση μέσω των συνομιλιών των έξι μερών που πρέπει να επαναληφθούν. Κάτι ακόμα που μας ενδιαφέρει είναι η κατάσταση ανθρωπιστική, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι ζωφερές. Υπάρχει συστηματική καταστολή και η Επιτροπή Έρευνας έχει καταδείξει ότι γίνονται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Χρειαζόμαστε πιο συγκεκριμένη διεθνή δράση για να σταματήσει η ατιμορρησία και να έρθουν ενώπιον τη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι. <clears throat> Θέλουμε επίση πιο στοχευμένε κυρώσει. Είναι απαραίτητο η διεθνή κοινότητα να πείσει την κυβέρνηση τη Κίνα να χρησιμοποιήσει την ε, επιρροή τη πολιτικά και οικονομικά για να υπάρξει αποκλιμάκωση στη χερσόνη τη Κορέα. Επίση, θα πρέπει να κάνει μια προσπάθεια να δεχτεί πρόσφυγε από τη Βόρεια Κορέα η κυβέρνηση τη Κίνα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Χέλμουτ Σόλτς έχει το λόγο από την ΓΚΟΕ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν συγκρούσεις και εξελίξεις στον κόσμο όπου κανείς αναρωτιέται αν υπάρχει αρκετή λογική στον κόσμο για να υπάρξει μια λύση. Η σύγκρουση στην Κορεατική Χερσόνησο είναι μια τέτοια περίπτωση για μένα υπάρχει όλη αυτή η ιστορική πορεία που οδηγεί σε σύγκρουση και ρητορική εχθρικού χαρακτήρα. Έχουμε συνέχεια ένα διάλογο ο οποίος είναι αντιπαραθέσεως και ο καθένας οχυρώνεται στις δικές του θέσεις. Στην περίπτωση Βόρειας Κορέας είναι σαφής, σαφές ότι υπάρχουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά και ο πόλεμος δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μια λύση ούτε ένα ρητορικό σχήμα. Ακόμα και σήμερα συνεχίζονται όλα αυτά. Μετά από την πρόσφατη καταδικαστέα πυρηνική δοκιμή <clears throat> της Βόρειας Κορέας, όλοι ε, μιλούν και ρητορεύουν, κανείς δεν δρά Γι' αυτό είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε σε, στην οδό που είχαμε αναφέρει στο ψήφισμα του 2013 και να, να επιμείνουμε στο θέμα των κυρώσεων. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει φύγει τόσο πολύ από την, από την επικαιρότητα το θέμα της Βόρειας Κορέας. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να αφήνουμε τη Βόρεια Κορέα να λειτουργεί χωρίς πραγματικές κυρώσεις. Με το να κάνουμε αυτή την διαδικασία δεν βλέπουμε ότι υπάρχουν τόσα πολλά iPhone τα οποία παράγονται στην Βόρεια Κορέα. Δεν μπορούμε φυσικά να μιλήσουμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν υπάρχει καμία μορφή δημοκρατίας στην ε, Βόρεια Κορέα. Υπάρχει βίαιη υποχρεωτική εργασία που απαιτείται από την ε, Βόρεια Κορέα και δεν μπορεί να υπάρχει καμία νομοποίηση σε μια τέτοια κεντρικά επιβαλόμενη δικτατορική οικονομία. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να κατευθυνθούμε προς την κατεύθυνση που έχει τονίσει το ψήφισμά μας και να ακολουθήσουμε μια νέα στρατηγική για να μπορέσει να επιληθεί η διαμάχη στην χερσόνησο της Κορέας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παντσέρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταδικάζουμε με τα στην πυρηνική δοκιμή που έκανε τον περασμένο Γενάρη στις 6 Ιανουαρίου δηλαδή η Βόρεια Κορέα και καλούμε το Βορρά να ε, ξαναεπιβεβαιώσει και να υπογράψει εκ νέου την Συμφωνία για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων από την οποία είχε αποσύρει την υπογραφή της το 2003. Χρειάζεται να να συμμορφωθεί με τις ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ η Βόρεια Κορέα διότι δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν επιτρέπεται την ύπαρξη αντιπολίτευση και το δικαστικό σύστημα ε, ελέγχεται από την κυβέρνηση. Ενώ οι νόμοι που ισχύουν θεωρούν αδικήματα ως, ε, κατά του κράτους οποιαδήποτε μορφή ελεύθερη έκδοση. θα έπρεπε η Βόρεια Κορέα να κληθεί ενώπιον του Διεθνού Δικαστηρίου για να ε, απαντήσει γιατί υπάρχουν τέτοιε παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Το ψήφισμα επίση ζητά την κατάργηση τη θανατική ποινή και την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων ώστε να μπορούν οι πολίτες να συνασπίζονται ελεύθερα ε, το ίδιο και για την στατικοποίηση της χώρας η οποία είναι ιδιαίτερα αυξημένη θα πρέπει λοιπόν να προβλεφθεί μέχρι και ανθρωπιστική βοήθεια για αυτή τη χώρα. Ευχαριστούμε κύριε Παντζέρη, μέρους του ΕΛΚ, η κυρία Σόντροπα. Για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κατάσταση στη Βόρεια Κορέα είναι πολύ δύσκολη. Την έπισκέφτηκα εγώ ίδια πριν από 10 χρόνια. Και είδα πραγματικά πως το καθεστώς φυλακίζει τους πολίτες και τους αναγκάζει να μείνουν, ζουν απομονωμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο. Από ό,τι φαίνεται και σύμφωνα με στοιχεία του 2014, ε, τίποτα δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 10 χρόνια. Ακόμη δεν είναι ελεύθεροι πολίτε στη χώρα, ενώ η κυβέρνηση χρηματοδοτεί τις πυρηνικέ δοκιμές και την ανάπτυξη τέτοιων όπλων, καθώς και την ε, οργάνωση δυνάμεων ασφαλείας που παρακολουθούν του πολίτε. Ο αφοπλισμός λοιπόν δεν υφίσταται και αυτό είναι πολύ κρίμα διότι η Βόρεια Κορέα είναι μια χώρα με τεράστιο δυναμικό που θα μπορούσε να είναι πολύ πλούσια ε, όπως η Νότια Κορέα και να προσφέρει αυτό το δυναμικό και στους πολίτες, τους, πολίτες της. Ε, δεν είναι στα χέρια όμως της Νότιας Κορέας η λύση. Θα πρέπει να έρθει από το απολυταρχικό ε, βορειοκορεατικό καθεστώς. Το Κοινοβούλιο παρακολουθεί στενά ε, το πώ ε, εξελίσσονται τα πράγματα στην Κορέα και κατανοεί πάρα πολύ καλά τι εξελίξει. Μετά το ψήφισμά μα, και εφόσον εγκριθεί, λέγεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλη τη την εμπειρογνωμοσύνη, καταρτίζοντα μια στρατηγική και για την Νότια Κορέα. Που και αυτή θα μπορούσε να συμβάλλει στην προσπάθεια. Εφόσον λοιπόν τα σύνορα τη Βόρεια Κορέα είναι κλειστά, θα πρέπει κάτι να κάνουμε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Ευχαριστούμε εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών η κυρία Κριστέα. Ο κύριος Κριστέα. Ευχαριστώ πολύ κύριε την Πρόεδρε. Η διάδοση πυρηνικών βιολογικών όπλων ε, απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια. Έξω και καταδικάζω ότι η πυρηνική δοκιμή που έκανε στις 6 Ιανουαρίου η Βόρεια Κορέα Πρόκειται για να παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας. Ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του Σύνδεξη για τη μηδιάδοση των ε, πυρηνικών όπλων. Όλες οι αστηριότητες ε, βαλιστικές ε, και οι διαδικασίες στο πλαίσιο του πυρηνικού προγράμματος πρέπει να διακοπούν άμεσα. Και θα πρέπει η χώρα να αναλάβει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ώστε να έχουν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις ε, και ο ειδικός επιστήμονας για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρόσβαση. Πρέπει να παραμείνουν οι διάβλοι επικοινωνία ε, και να ισχύσουν ε, τα ανθρωπιστικά προγράμματα, αλλά οι βορειοκορετικές αρχές θα πρέπει να παρέχουν τροφή σε όλους τους πολίτες και να τους εξασφαλίζουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Λυπούμε, αλλά πρέπει να διακόψω για δύο λεπτά την ε, συνεδρία. Σε Ευχαριστώ. I'm sorry. On behalf of the group. Σας ζητώ συγγνώμη. Κύριε Στέμεσβάκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να είστε καλύτερα. Η Βόρεια Κορέα πριν από δύο εβδομάδες με, το, με τη δοκιμασία θερμοπυρηνικών, ε, θερμοπυρηνικής βόμβας δημιουργήσαν μεγάλη ανησυχία στον κόσμο. Είναι μια ζωφερή χώρα η Βόρεια Κορέα. Όλα αυτά τα οποία ξέρουμε είναι ότι οι άνθρωποι εκεί ζουν σαν σκλάβοι και υπάρχουν συνεχιζόμενε παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κανεί δεν έχει την ελευθερία τη γνώμη του. Οι πολιτικοί ηγέτε αντιπολίτευση έχουν φρικτό τέλο. Υπάρχει καταναγκαστική εργασία, ε, ο κόσμος πεθαίνει από την πείνα. Το πείραμα αυτό λοιπόν έγινε με τη βοήθεια της Ρωσίας και της Κίνας που είναι σύμμαχοί του, αλλά κανείς δεν αναφέρθηκε σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν μπορεί να παραμείνει σιωπηλή. Έχουμε καθήκον στις εκατοντάδες χιλιάδες αθώων ανθρώπων που είναι χωρίς ε, τροφή, χωρίς ε, μέλλον για όλη τη γενιά της Βόρειας Κορέας που θα πρέπει να ζήσει σε αυτές τις κατάστασεις. Κυρία Χαρατσόβα, από την ομάδα των Φιλελευθέρων έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Η Βόρεια Κορέα εξακολουθεί να είναι κάτι το κατεπήγον. Κάθε μήνα έχουμε νέες ειδήσει για κάποιο άτομο το οποίο φυλακίζεται αδίκως και για κάποια εκτέλεση κάποιου κυβερνητικού αξιωματούχου οι ακόμα περισσότεροι πολίτες Βόρειας Κορέας πεθαίνουν από την πείνα για να τροφοδοτήσουν μια στρατιωτική μηχανή. Το να πούμε ότι είναι μια καυκική <clears throat> χώρα η Βόρεια Κορέα δεν αποδίδει την πραγματικότητα. Μετά από την πυρηνική δοκιμή των προηγουμένων εβδομάδων τώρα λένε ότι βρήκαν έναν τρόπο για να ξεπερνάνε τον πονοκέφαλο μετά από μεθύση. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι μας οδηγούν στο συμπέρασμα δεν μπορούμε να ζητήσουμε τίποτα από την κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας. Μόνο μπορούμε να ζητήσουμε από την Κίνα να σταματήσει την υποστήριξή της για την Βόρεια Κορέα που οδηγεί σε κατασπατάληση φυσικών πόρων, χρημάτων <clears throat> και είναι ένα όνειδος για τους Κινέζους. Έχει τελειώσει ο, πικρό, ο πόλεμος. Η υποστήριξη αυτής της κυβέρνησης δεν βοηθάει καν την κινέζικη ασφάλεια. Μόνο μια ενωμένη Κορέα μπορεί να φέρει πραγματική ασφάλεια στη Βόρειο Ανατολική Ασία. Ευχαριστώ. Από την ομάδα EFTT ο κύριος Άρνοτ. Ένα λεπτό παρακαλώ. Όπως όλες οι λαϊκές δημοκρατίες, η Βόρεια Κορέα δεν είναι λαϊκή, δεν είναι δημοκρατική και δεν κάνει τίποτα για το λαό της. Ο κομμουνισμός στη Βόρεια Κορέα, όπως και όλα τα άλλα τέτοια καθεστώτα, είναι σάπιος και διεφθαρμένος. Κάθε τέσσερις ώρες εκτελούν κάποιον χρησιμοποιούν πιο πολλά ναρκωτικά από τη τρόφιμα. Όλα με το κουπόνι και χρησιμοποιούν τρομερή βία κατά των αντιφρονούντων. Λυπάμαι, αλλά πριν από λίγους, από δύο μήνες στο Βρετανικό Κοινοβούλιο ο Σκιώδης ε, οικονομικός, Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στο μικρό κόκκινο βιβλίο του Μεγάλου Τιμονιέρ. Αλλά και αυτός οδήγησε στο θάνατο δεκάδες εκατομμυρίων ανθρώπων θα πρέπει να νιώθουμε ντροπή που υπήρξε ποτέ τέτοιο εξτρεμισμό στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να απορρίψουμε την πολιτική τη Βόρεια Κορέα, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ιδεολογία αυτή και θα πρέπει να σταματήσουμε αυτό που κάνουν οργανισμοί τρομοκρατικοί όπως η Βόρεια Κορέα και η ISIS. Ο Νικολά Μπαΐ έχει το λόγο. Στην παράγραφο 3, στο κοινό ψήφισμα, λέτε ότι θυμείτε την εξέβρεση διπλωματικής λύση με την πηγιόν Γιάνγκα, αλλά στην επόμενη παράγραφο απαιτούνται νέε κυρώσει, Ενώ η Βόρεια Κορέα ήδη είναι η πιο απομονωμένη χώρα στον πλανήτη. Φυσικά και δεν έχω καμία συμπάθεια στην τερα... τρομερή αυτή κομμουνιστική δικτατορία, αλλά δεν νομίζω ότι στις προκλήσει πρέπει να απαντάμε με νέε ε, κυρώσει, γιατί αυτή την παράνοια θα την ε, εξα... Ε, οξύνουμε ακόμη περισσότερο. Πρέπει να δούμε και τι κάνουν ε, ε, οι δυτικές χώρες που πολλές φορές δίνουν ε, πιστικά επιχειρήματα σε αυτούς τους παρά. Ξέρουμε τι έγινε με το πρόσχημα για το δεύτερο πόλεμο του κόλπου και που ευθύνεται για την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η όλη περιοχή δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει συνέχεια να αναμειγνύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πολλές φορές έτσι οξύνει αντί να μετριάζει τις συγκρούσεις εκεί. Θα πρέπει λοιπόν να, να από τη Βόρεια Κορέα να βρει λύση στα πραγματικά προβλήματα που την ταλανίζουν. Ευχαριστώ. Ο κ. Τζουλίτσα έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου προς το σχέδιο ψηφίσματος που καταδικάζει στεναρά την πυρηνική δοκιμή που έκανε στις 6 Ιανουαρίου 2016 η Βόρεια Κορέα. Μία ακόμη πυρηνική δοκιμή από τη χώρα αυτή που για μια ακόμη φορά ε, μας δείχνει ότι πρόκειται για μια απειλή για την ε, ασφάλεια και την ειρήνη στον πλανήτη. Υπάρχουν ψηφίσματα του ΟΗΕ μιλούν για το παράνομο βαλιστικό πρόγραμμα και παράνομο πυρηνικό πρόγραμμα που καταπατούν τις διατάξεις των αστικών περίμη πυρηνικών όπλων ε, και ε, δημιουργούν περισσότερες εντάσεις με την πολιτική όπλων βασικής καταστροφής ε, δεν κάνει καλό δεν, η χώρα αυτή ούτε στους πολίτες. Πρέπει να επανέλθει στον διάλογο των έξι. Περιμένω ενίσχυση των κυρώσεων από το Συμβούλιο Ασφαλείας το ε. και καλό την Βόρεια Κορέα τελικά να επιλέξει ε, το επικοδομητικό ε, μονοπάτι. Ευχαριστώ. Ωραία για τη διαδικασία Catch the Eye. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ στηρίζω το ψήφισμα αυτό. Επιτέλους η Βορεια Κορέα πρέπει να, είναι μια χώρα που θα την αντιμετωπίσουμε ως χώρα που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι μια κομμουνιστική δικτατορία που οδηγεί στην πείνα εκατομμύρια πολίτες είναι 15% του πληθυσμού που ζουν κατά το κατόφλι της φτώχειας, υποσυτίζονται και πεθαίνουν. Θα πρέπει λοιπόν να αναθερμανθεί ο διεθνή διάλογο για τη χώρα αυτή και είναι πραγματικά άριστη η κίνηση να υιοθετήσουμε αυτό το ψηφίσμα σήμερα. Θα πρέπει να ε, καλέσουμε την Κίνα να μας βοηθήσει στην όλη προσπάθεια, να ασκήσουμε πίεση στη Βόρεια Κορέα. Η Κίνα είναι η μόνη χώρα με κάποιο κύρος που θα μπορούσε, θα μπορούσε να ε, αλλάξει, να βοηθήσει να αλλάξει το καθεστώς στη Βόρεια Κορέα και να γίνουν σεβαστά στα θεμελιώδη ε, δικαιώματα. Ευχαριστούμε ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Βόρεια Κορέα παραμένει μεταξύ των ε, χωρών του κόσμου που προκαλούν με τις πυρηνικές δοκιμές και την βόμβα υδρογόνου που έκανε τον περασμένο Ιανουάριο. Είναι πολύ εύκολο βεβαίως να καταγγέλουμε την ε, συμπεριφορά της Βόρειας Κορέας γενικότερα. Τώρα ο κίνδυνος είναι πραγματικός. Πρόκειται για την τρίτη πυρηνική δοκιμή της Βόρειας Κορέας που οδήγησε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ να εγκρίνει νέες κυρώσεις κατά της χώρας αυτής. Ε, ήδη προστέθηκαν στις προηγούμενες οι νέες Η Βόρεια Κορέα δεν θα πρέπει να περάσει σε νέες πράξεις και ενέργειες πρόκλησης, σεβόμενοι τις διεθνείς της υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. Ταυτόχρονα η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να υιοθετήσει συγκεκριμένα μέτρα για να θέσει τέρμα στην κατάσταση αυτή. Οι μεγαλύτεροι παράγοντες, ε, όπως η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας, παγκοσμίω θα πρέπει να ασκήσουν την ε, πίεση και την επίδρασή του στην κυβέρνηση τη Βορεια Κορέα, ώστε να βεβαιωθούμε ότι η κατάσταση δεν θα υποβαθμιστεί έτσι περαιτέρω. Θα πρέπει να δούμε την Κορέα ως την τελευταία χώρα που έχει τέτοιο μεγάλο πρόβλημα παγκοσμίω. Ευχαριστούμε. Μάριο Πίντο. Η Βόρεια Κορέα μπορεί να αντιμετωπιστεί με τρόπο μόνιμο εάν η λύση ευρεθεί σε ένα πολυμερές πλαίσιο. Δεν μπορεί να είναι μονάχα η Ευρωπαϊκή Ένωση οι Ηνωμένε Πολιτείε μαζί με την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα που θα επιτύχουν κάτι τέτοιο. Πρέπει να συμμετάσχουν όλες οι χώρες που μπορούν να δώσουν με αυτό, συγκεκριμένα η Κίνα και η Ρωσία, που στο παρελθόν υπήρξαν σημαντικοί σύμμαχοι της Βόρειας Κορέας. Το να γνωρίσουμε λοιπόν την Κίνα και τη Ρωσία ή να τις γελιογραφούμε δεν οδηγεί σε μια λύση του προβλήματος, μπορεί απλώς να το επιδεινώσει. Το πρόβλημα των πυρηνικών εξοπλισμών της Βόρειας Κόρεας δεν θα λυθεί με ρητορικέ δηλώσεις. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες ενέργειες. Ευχαριστώ. Στετινά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, θέλω να τονίσω ότι στη Βόρειο Κορέα παραβιάσεις ανθρωπινών δικαιωμάτων διαπράττονται από ένα κομμουνιστικό καθεστώς, το οποίο απειλεί όχι μόνο την κορεατική χερσόνησο, αλλά και το μέλλον της δημοκρατίας στον κόσμο και στην Ευρώπη. σα προειδοποιώ. Προσπαθούν να διεθνοποιήσουν τον κομμουνισμό εκ νέου οι κομμουνιστές. Έχουμε το κόμμα στην Βοημία Μοραβία. Ο επικεφαλής της είναι ο πρωτεργάτης αυτού του νέου κινήματος. Προσπαθεί να δημιουργήσει μια νέα κομμουνιστική διεθνή. Με ισχυρό σύμμαχο τους κομμουνιστές από τη Βόρεια Κορέα. Που συχνά πυκνά συμμετέχουν στις συνεδριάσεις που γίνονται στην Πράγα. Ευχαριστώ. Κύριος Ράντος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η Βορεια Κορέα είναι μια χώρα που έχει υπογράψει τις περισσότερες συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι οποίε βέβαια παραβιάζει ε, συχνά πυκνά. Πρέπει λοιπόν να σεβαστεί τα ε, ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλής όπως ζητούμε, καθώς και το Διεθνές Δίκαιο. Δεν βοηθάνε όμως οι εκκλήσεις στην προκειμένη περίπτωση. Και δυστυχώς ούτε και αν η Κίνα ασκήσει την επιρροή της στη Βόρεια Κορέα θα βοηθήσει. Γιατί αυτό θα το κάνει για να προωθήσει τα δικά τη συμφέροντα. Η μόνη λοιπόν λύση είναι με μια συντονισμένη διεθνή δράση. Κάτι το οποίο λείπει αυτή τη στιγμή. Διότι οι χώρες ε, γειτονικέ ε, δυσκολεύονται να συμφωνήσουν μεταξύ του. Παρ' όλα αυτά στηρίζω το ψήφισμα και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακολουθούν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα και τις προσπάθειές της να ε, αποσταθεροποιήσει τον πλανήτη. Η κυρία Κριστίνα Μορβάη, η επόμενη μιλητρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ελπίζω να αισθανθείτε καλύτερα πολύ γρήγορα. Στο σημείο 4 της έκθεσης ε, γίνεται λόγος για το Ευρωκοινοβούλιο που καλεί τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση για να πάψει η ατιμορρησία των δραστών και υπενθυμίζει ότι πρέπει να λογοδοτήσουν για τις μέχρι τώρα πράξεις τους που έχουν παραμείνει ατιμόρυτες. Κύριε Επίτροπε, σωστά θυμάμαι, υπάρχει μια πληθώρα πρώην κομμουνιστικών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την αρχή των διαπραγματεύσεων για την διεύρυνση, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων προσχώρησης και Εφ' κάλεσε ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση τις χώρες της ένταξης να φέρουν τους δράστες αυτών των ε, απεχθών εγκλημάτων ενώπιον της δικαιοσύνης. Θυμάμαι σωστά ή λάθος. Ή πάλι μιλάμε για διπλά μέτρα και σταθμά. Ευχαριστώ. Πάετ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, δεν θα μπορούμε να συζητάμε στα κατεπήγοντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα τη Βόρεια Κορέα κάθε φορά. Είναι πράγματι ένα πολύπλοκο πρόβλημα και ιδίως για το λαό της ε, Βορείου Κορέας. Είναι φανερό ότι ο κίνδυνος όμως της Βόρειας Κορέας γίνεται όλο και μεγαλύτερος για τις όμορες χώρες. Μπορούμε να διδαχτούμε από την ιστορία που μας λέει ότι αν είχαμε παρέμβει εγκαίρως πολλά προβλήματα θα μπορούσαν να είχαν ε, εμποδιστεί. Και η Βόρεια Κορέα είναι μια τέτοια περίπτωση. Μιλάμε για τη Βόρεια Κορέα. Αλλά οι χώρες που μπορούν να ασκήσουν πίεση αυτή τη στιγμή δεν κάνουν τίποτα. Μιλάμε για τη Ρωσία και την Κίνα. Όλοι πρέπει να μάθουμε λοιπόν από τα σφάλματα του παρελθόντος. δεν πρέπει να αφήσουμε την κατάσταση να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ρίκιο και ο επίτροπο Επίτροπος Μιμίτσα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη λαοκρατική δημοκρατία της Βόρειας Κορέας, όπως μεταξύ άλλων ε, τεκμεριών και η έκθεση ε, στις αρχές του 2014. Η κατάσταση είναι κατεπίγουσα και απαιτεί συστηματικές ε, διαρθρωτικές αλλαγές στη Βόρεια Πρόκειται για ηθική ε, επιτακτική ανάγκη, πολιτική επιτακτική ανάγκη, είναι όμως και κατεπήγον γιατί η κατάσταση αυτή είναι συνταγή για μακροχρόνια ε, περιφερειακή αστάθεια. Υπενθυμίζω ότι ορισμένα από τα πορίσματα αυτής της Κριστασικής Επιτροπής ε, ε, καταδεικνύουν μέχρι και το ενδεχόμενο ε, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τη σύσταση το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να παραπέμψει την κατάσταση στην Βόρεια Κορέα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε και θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή αυτό που προσπαθούν να, να παραμείνει στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας κατά προτεραιότητα σε αυτή την δινή κατάσταση. Όμως, ο στόχος Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι απλά τα πρωτοσέλιδα ή οι καταγγελίες. Ο βασικός πρωταρχικός μας στόχος είναι η επίτευξη σημαντικών βελτιώσεων επιτόπου και σημαντικής πρόοδου, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη χρηματοδοτεί προγράμματα επιστηστικής βοήθειας, σύντρευσης, αποχέτευσης στην ελλακρατική Δημοκρατία της Βόρειας ε, Κορέας. Θα βοηθήσουν σημαντικά τον ενδύπληθισμό και παιδιά που βρίσκονται σε διάφορα ε, ιδρύματα ή τους ηλικιωμένου ή άτομα με αναπηρία ή αγρότες, ευάλωτους κτλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να κάνει πιο πολλά ακόμη, να συνεργαστεί ακόμη περισσότερο με τις αρχές της ε, Βόρειας Κορέας, μόνο όμως όταν η χώρα αυτή με αξιόπιστο ε, και ουσιώδη τρόπο αντιμετωπίσει ε, τι σοβαρέ ανεπαρκίε τη ε, στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αν αποφασίσει η Βόρεια Κορέα να ακολουθήσει ε, το δρόμο τη πραγματική δέσμευση και προσήλωση στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αρχίζοντα από το να συνεργάζεται πλήρω με του μηχανισμού ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, τότε πραγματικά θα εξασφαλίσει ε, την ασφάλεια ε, και θα μας καθησυχάσει στο ότι δεν θα δημιουργήσει ποτέ παράνομα πυρηνικά όπλα. Οι πρόσφατες όμως ενέργειες της Βορείου Κορέα με την παράνομη πυρηνική δοκιμή, την οποία εξήγαγε στις 6 Ιανουαρίου, δείχνουν ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο δεν έχουμε κάποια θετική εξέλιξη. Είναι πολύ λίγες οι δυνατότητες συνεργασίας με τη χώρα αυτή ω εκ τούτου. Θα πρέπει η Βόρεια Κορέα να εστιάσει στις αναγκαίε μεταρρυθμίσει στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν θα πρέπει να αποσταθεροποιεί, ούτε να προβαίνει σε παράνομες ενέργειες που δημιουργούν ένα σταθές και επικίνδυνο περιβάλλον σε βάρος όλων. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Έχω λάβει 7 προτάσεις ψηφί.